Einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Mitglieder. Καλημέρα συνάδελφοι. Βλέπω ότι έχετε προσέλθει μαζικός. Είναι και ψηφοφορία σήμερα. Ξέρω επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ε, θα έλεγα να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. Καλημέρα, ξαναλέω. Sie sehen, ich spreche Deutsch. Alle <laughs> haben die Μιλάω γερμανικά. Καλώς βάλατε τα ακουστικά σας. Ξεκινάω λοιπόν. Στα μέλη της Επιτροπής. Περνάμε ευθύς αμέσως στην ημερήσια διάταξη της σημερινή συνδυράσης. Αν δεν υπάρχουν ε, προτάσεις αλλαγή τροποποίησης, θεωρείτε ότι εγκρίνεται. Και να περάσω ευθύ αμέσω ε, στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Στις 30 Σεπτεμβρίου Μέσω γραπτής διαδικασίας, μεταξύ 7 και 18 Οκτωβρίου, οι συντονιστές αποφάσισαν τα εξής. Εξοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων ε, ιδίας για τα εξή θέματα. Υπέρβαση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, συμμετοχή γυναικών στην ψηφιακή οικονομία. Δεύτερον, κατάσταση όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών. Τρίτο θέμα. Προώθηση της ισότητας των φύλων στην επιστήμη, στα επαγγέλματα, στην ε, τεχνολογία, στην μηχανική και στα μαθηματικά, στην εκπαίδευση και στις ε, επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Τέταρτον, ισότητα ε, φύλων στον ε, τομέα της εξωτερική πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτον, αντίκτυπος ε, της ενδοοικογενειακή βίας στις γυναίκες και στα παιδιά και έκθεση παρακολούθησης με θέμα ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και μια έκθεση ιδία πρωτοβουλία νομοθετικού χαρακτήρα με θέμα την αντιμετώπιση της βίας εναντίον των γυναικών στο διαδίκτυο και μια έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία ε, που αφορά την διακίνηση ανθρώπων. Επόμενο θέμα, επόμενη απόφαση των συντονιστών. Σύνταξη προφορικού, προφορικής ερώτησης όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Ανάθεση έκθεση ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων στην ε, ομάδα των Σοσιαλιστών ορισμός της κυρίας ε, Τολερέ και της κυρίας Δελβός Κόρφιλτ ως ε, μονίμων συνεισηγητριών για την συμπερίληψη της διάστασης του φίλου. Εξοδότηση προγράμματος ακροάσεων και αποστολών για το πρώτο εξάμεινο του 20 και πρόγραμμα επερχόμενων μελετών και εργαστηρίων και αποφασίστηκε επίσης σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις να γίνει ε, συνάντηση και συζήτηση με την γαλλομαροκινή ε, δημοσιογράφο Λέιλα Σλιμάνη. Αυτά. Ε, εμείς ξεκινάμε, ακόμη και αν δεν έχει ακόμη ξεκινήσει το σχετικό έργο η Κομισιόν, το δικό μας έργο για να μπορέσουμε να είμαστε και έτοιμοι όταν ξεκινήσει η Κομισιόν. Θέλω επίσης να σας επισημάνω από πλευράς μου το εξή. Υπάρχει ένα email το οποίο έχετε λάβει και θα το ξαναλάβετε από μια καλλιτέχνηδα η οποία ε, πραγματοποιεί έκθεση εδώ στις Βρυξέλλες στο Δεκέμβριο. Εργάζεται σε ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό project και θα σας, απευθύνει, θα σας απευθυνθεί για να σας μιλήσει και να σας φωτογραφίσει ενδεχομένως. Σας, το, σας ευχαριστώ την προσοχή, γιατί πραγματικά είναι μια καλλιτέχνητα εξαιρετικά άξια ε, να μην καταλήξει το email αυτό κάπου στον ε, φάκελο με τα ανεπιθύμητά σας. Δώστε του την απαραίτητη προσοχή. Περνάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες τώρα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Ετήσια έκθεση για το 2018. Δεν είναι πολύ μακρύς ο κατάλογος ε, της ψηφοφορία. Ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε περίπλοκα θέματα, αν και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα για κατατιμήματα ψηφοφορίας, οπότε θα ήθελα να έχετε έτοιμες τις ε, ε, κάρτες ψηφοφορίας σας. Δεν θα τις ε, χρησιμοποιούμε συνεχώς, όμως ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να επαληθεύσουμε. Οπότε ξεκινάμε με τη γνωμοδότηση αυτή. Ε, παράγραφος 1. Ε, κατά τμήματα ψηφοφορία. Οπότε ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ας μην το κάνουμε ηλεκτρονικά, ας το κάνουμε διανατάσσεω ισχυρό και μετά αν υπάρξει πρόβλημα θα το επαληθεύσουμε. Παράγραφος 1, σοφορία κατά τμήματα για το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα για την παράγραφο 1, υπέρ. Κατά. Αποχές επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Της ε, παραγράφου 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Κατά τμήματα πάλι. Πρώτο τμήμα. Υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. zum 3. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στο τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα.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 Και τώρα περνάμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα, ηλεκτρονικά, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 ψηφίπερ, 6 κατά, μία αποχή. Σαφές το αποτέλεσμα. Και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων το σχετικό προφορικό ερώτημα. Παράγραφος 4, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και Τέταρτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε ξανά σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κείμενο της προφορικής ερώτησης ε, στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία, 24 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια. Damit sind die Abstimmungen beendet. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Στα επόμενα σημεία, 6-7, απαλλαγή 2018, Έχουμε συντάξει δύο γνωμοδοτήσει για την ε, Επιτροπή Προπολογισμών. Η μία αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ισότητα των Φύλων και το άλλο αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ο, η συντάκτρια των γνωμοδοτήσεων ε, η Φράνσις ε, Φιτζέλατς πρότεινε να τις δούμε μαζί αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τις δύο αυτές προτάσεις. Σας ευχαριστώ που δέχεστε να τις δούμε μαζί. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω στους συναδέλφους ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 8 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Οπότε υπάρχει ακόμα δυνατότητα υποβολής για αλλαγέ. Ε, χαίρομαι που μπορώ να παρουσιάσω λοιπόν δύο διαφορετικά αλλά αλληλένδετα. Με συγχωρείτε, εάν μπορείτε, τα ακουστικά σας για να μην έχουμε παρεμβολές. Ναι, ε, έχουμε λοιπόν τις δύο αυτές αλληλένδετες εκθέσεις σήμερα. Την απαλλαγή του 2018 για το ΕΙΓΕ, e το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γενικό Προπολογισμό. Τις εκθέσεις αυτές τις βλέπει έτσι η Επιτροπή Ελέγχων του Προπολογισμού. Η απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επικεντρώνονται κυρίως στα θέματα ευθυγράμμισης της διάστασης του φύλου για την προστασία και την αξιολόγηση της υλοποίησης που είναι πολύ σημαντική. Επίση, θέλουμε να γίνει η ανάλυση, η λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων και όχι απλώ η ε, συνάθρησή τους για του 27 τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για συγκεκριμένα προγράμματα. Τώρα για τα διαφορετικά μεμονωμένα προγράμματα χρειάζεται δημοσιονομική γραμμή ανάλογα με το στόχο που προβλέπεται στα πλαίσια του προγράμματος για την ισότητα και την ιδιότητα του πολίτη και αναγνωρίζεται η σημασία του, πολιτικού, του πολιτικού προγράμματος βάσει των δεδομένων που θα πρέπει μάλλον να χρησιμοποιούν δεδομένα και για, για το θέμα της έμφυλης βίας. Επαναλαμβάνουμε το αίτημα, ε, κάθε στόχο στα πλαίσια του προγράμματος, ε, στη συγκεκριμένη διάσταση τη ισότητα των φύλων, να ελέγχεται και να υπάρχει και λογοδοσία. Η έκθεση τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη έμφαση στην προοπτική της διάστασης των ε, φύλων και της ισοσοδητάς τους και στο Horizon 2020 και στο θέμα της καινοτομία. Επειδή δίνεται μεγάλη έμφαση στον προπολογισμό στο θέμα αυτό, θα πρέπει και αυτό να συμβεί. Επίσης, σε ό,τι αφορά την έκθεση για το ΕΕΚΕ, Καλωσορίζουμε την, εργασία, της εργασίας, την καλή δουλειά του Ινστιτούτου μέχρι τώρα. Καλωσορίζουμε την στρατηγική για την διαχείριση των γνώσεων ε, και την επικοινωνιακή τους πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και την αντιμετώπιση της βίας στο χώρο εργασίας και τη συνεργασία με τα εθνικά δίκτυα και μία επαφής. Νομίζω ότι η εκτέλεση του προπολογισμού τους υπήρξε άριστη ως τώρα με βελτιώσεις που είναι δυνατές και στο επίπεδο των δεσμεύσεων και στο επίπεδο των ε, ε, δαπανών. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο δίνει κάποιε ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν νομικές και γενικέ βελτιώσεις και νομίζω ότι μπορούμε να συστήσουμε στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών από την προοπτική της δικής μας της επιτροπή να δώσει την απαλλαγή στο Διευθυντή του ΕΚΕ ε, ε, για την ε, εκτέλεση του προπολογισμού το 2018. Ευχαριστώ την Γραμματεία για τη σύνταξη των δύο αυτών εκθέσεων και όπω είπα, εάν υπάρχουν τροπολογίες σημεία τα οποία ενδεχομένω οι συνέδελφοι θα ήθελαν να ε, παρατηρήσουν. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ, Βίλια. Με ευχαριστώ. Είμαι ισχυώδης εισηγήτρια των σοσιαλιστών. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την συνάδελφο Φράνσις Φιτζεράλτ για το σχέδιο έκθεσης για το ΕΓΚΕ και την απαλλαγή του 2018. Δεν έχω πολλά να προσθέσω διότι το σχέδιο πραγματικά επικεντρώνεται σε πολύ σοβαρά σημεία. Δεν είχαμε προβλήματα με την εκτέλεση του προπολογισμού του ΕΚΕ. Πραγματικά το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων είναι σοβαρός παράγοντας για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι τώρα είχαμε άριστη συνεργασία από την ε, ίδρυσή του και μετά η δουλειά του ΕΚΕ είναι μεγάλη σημασία σας προ την ανάλυση των δεδομένων που πρέπει να είναι άρεστη ποιότητα και να οδηγήσουν και στι ανάλογε μελέτε. Πολύ σημαντικό υλικό για τη δική μα τη δουλειά. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ, Φράνση. Προφανώ συνεργαστήκαμε για το σχέδιο αυτό γνωμοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για το σχέδιο γνωμοδότηση για το Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ μερικές γενικές παρατηρήσεις. Η γενική ευθυγράμμιση του θέματος της διάστασης των ε, φύλων και της ισότητας των φύλων πρέπει να γίνεται σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις διέπει όλες και αυτό είναι κυρίως ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα αν μιλάμε για την δημοσιονομική διαδικασία θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών ταυτόχρονα και στην υλοποίηση του προπολογισμού και στην αξιολόγηση της υλοποίησης. Χρειάζονται σίγουρα περισσότερες στοχευμένες δράσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων και συγκεκριμένες δημοσιονομικές γραμμές για τους ε, αντίστοιχους σκοπούς. Δεν είναι αποδεκτό το πρόγραμμα Δάφνα να μην έχει συγκεκριμένη δημοσιονομική γραμμή. Είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ κακό που μειώθηκε για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο το, το σχετικό ποσό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ανανεωμένη δέσμευση από όλα τα θεσμικά όργανα και να υπάρξει συμφωνία για μια στρατηγική ισότητα των φύλων με συγκεκριμένη μέτρηση των στόχων, με στοχευμένες δράσεις και τα ανάλογα ποσά στον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την ε, κύριο εισηγήτρια και θα συνεργαστούμε ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να βελτιωθεί το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστούμε. Δεν είστε απλώ μια και εισηγήτρια, αλλά και πρώην πρόεδρο τη ε, Επιτροπή ε, των Δικαιωμάτων των Γυναικών και γνωρίζετε καλά τα θέματα του ΕΙΓΕ. Θα μιλήσω εξ ονόματο των ε, Πρασίνων. Θα ήθελα να πω ότι καλώς ορίζουμε και αποδεχόμαστε είναι την έκθεση <clears throat> για την απαλλαγή όσον αφορά το Ινστιτούτο Ισότητας φίλων για το έτος 2018. Εδώ παίρνω το λόγο εξ ονόματος της κυρίας Μόνικα Βένελ που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και η οποία εργάστηκε ε, για το ε, θέμα ε, του Ινστιτούτου Ισότητας Φύλων ασχολήθηκε δε και με τα διορθωτικά ταμεία και με τη γενική εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2019 ήδη αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, περισσότερη πρόοδος όσον αφορά τη συνεκτίμηση ε, της διάστασης ε, φύλου. Μόναχα ένα ε, ε, βαθμό, κατά μία μονάδα αυξήθηκε ε, η χρηματοδότηση θεμάτων που αφορούν τη διάσταση φύλου το προηγούμενο έτος. Οι πληροφορίες που δίνονται από το Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων είναι θεμελιώδου σημασίας για την Επιτροπή μας. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε την απαλλαγή και να ζητήσουμε και από την Επιτροπή Προϋπολογισμού να υπάρξει πλήρη συνεκτίμηση της διάστασης ε, του φύλου σε όλες ε, τις ε, δραστηριότητες. Το Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για την ισότητα. Όσον αφορά το γενικότερο θέμα της απαλλαγής για τους, για τους οργανισμούς κλπ για το οικονομικό έτος 18, Επιτροπή και Εκτελεστικοί Οργανισμοί, ε, ε, η ομάδα μου θα υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες. Όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να δεσμευτούν για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου. Επίσης, είναι κρίμα που βάσει της ψηφοφορίας δεν έγιναν σοβαρά βήματα για τον προπολογισμό του 20 ε, και επίσης ε, η Κομισιόν θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη τα στοιχεία αυτά. Τρίτον, ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι έτσι ώστε να προωθηθεί το θέμα της ισότητας των φύλων. Ε, δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώνει διαρκώς τους πόρους που ε, δίνει για την ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και κατά αυτή την έννοια το πρόγραμμα Δάφνη θα πρέπει να συνεχιστεί με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη τα οικονομικά αλλά κοινωνικά και οικολογικά ε, ε, στοιχεία και προϋποθέσεις στην συνεκτίμηση και του αντικτύπου των μέτρων όσον αφορά τη ισότητα των φύλων πριν αυτά εγκριθούν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται μία gender budgeting ρήτρα σε όλες τις συμφωνίες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόμενη ομιλήτρια. Θα ήθελα με δύο λόγια να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την τεράστια δουλειά που έκανε όσον αφορά την απαλλαγή για το 2018, κυρίως δεν την απαλλαγή για το Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων. Ε, εμείς θα θέλαμε όντως να υπάρχει gender budgeting δηλαδή στην εκτίμηση τη φύλου στην κατάρτιση του προπολογισμού. Ε, και αυτό μπορεί να γίνει έγκαιρα μονάχα εάν έχουμε στη διάθεσή μας τους δείκτε αυτούς που θα μας επιτρέψουν να ε, μετρήσουμε την πρόοδο που ε, μπορεί να έχει γίνει σε κάθε επίπεδο. Και βεβαίως ο ρόλος του Ινστιτούτου Ισότητας φύλων ε, σε σχέση και με του, τις προβλέψεις του ΠΔΠ θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ε, που να διασφαλίζει ότι οδηγούμεθα προς αυτήν την ισότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η Κριστίνα Άντερσον. Äh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, γνωμοδότηση αυτή. Δυστυχώς στα social media τις τελευταίες εβδομάδες ε, εμφανίστηκαν πολλές γυναίκες οι οποίες διαμαρτύρονται ε, ότι το Ινστιτούτο αυτό δεν εξασφάλισε τα ίσα δικαιώματά τους όσον αφορά τα μισολογικά ζητήματα, τα εργασιακά ζητήματα ε, που συχνά πρόκειται για γυναίκες που εργάζονται μέσω προκτορίων εργαζομένων και γι' αυτό προτιμώνται και από αυτέ τι εταιρείε. Σω λοιπόν η Επιτροπή μα θα πρέπει να ασχοληθεί και με αυτό το θέμα. Δεύτερο ερώτημα. Είχαμε εδώ μια εμπειρογνώμονα που ξεχνάω δυστυχώ το όνομά τη. Πάντως ε, μας είχε ενημερώσει σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και είχε εκφράσει τότε ε, την ε, δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία μόλις μέχρι το 2012. Υπάρχουν πληροφορίες γιατί συμβαίνει αυτό, υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Αν όχι γιατί, μήπως ε, οφείλεται σε προβλήματα χρηματοδότησης του Ινστιτούτου, μήπως υπάρχουν ζητήματα οικονομικά τα οποία δεν επιτρέπουν στο Ινστιτούτο να συλλέγει τέτοιου είδους δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση να το, δια, να το διαρευνήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, αυτό, αυτά είναι ερωτήματα που δεν απευθύνονται βεβαίω μόνο στην εισηγήτρια στην οποία θα δώσω ε, το λόγο, αλλά απευθύνονταν και σε μένα. Γι' αυτό και θα απαντήσω εντάχει. Στις 5 Δεκεμβρίου ε, θα έχουμε εδώ μαζί μας την ε, πρόεδρο του ΕΙΓΕ και βεβαίως ε, με χαρά θα απαντήσει στα ερωτήματα που ε, θέσατε εσείς. Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, εντός της προθεσμίας μπορείτε βεβαίως να υποβάλλετε και ε, τις σχετικές τροπολογίες. Ίσως θα ήθελε και η συγγήτρια βεβαίως να τοποθετηθεί για τα όσα ακούστηκαν, τα σχόλια των συναδέλφων. Παρακαλώ, συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, Εύλην. Νομίζω ότι είναι σαφές από τα όσα είπαν οι συνάδελφοι και σας ευχαριστώ πολύ για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των σχολείων ε, ότι σκοπός μας πρέπει να είναι να τονίσουμε και να αναπτύξουμε ε, το, τη σημασία της συμπερίληψης της διάστασης του φύλου. Και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε και κάποιους τομείς στους οποίους θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει. Θα λάβουμε λοιπόν τις ε, τροπολογίες σας Έω την ημερομηνία που έχει προθεσμία. Νομίζω όμως ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα συμφωνήσουμε, γιατί αυτό που θέλουμε όλοι είναι να ενισχύσουμε ε, αυτό το ζήτημα και θα το κάνουμε μέσω της ε, έκθεσης, ε, γιατί είναι πραγματικά κρίσιμη και η περίοδος εν ώψη και της κατάρτισης του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου να υπάρχει έντονη διάσταση του φύλου και στην κατάρτιση του προπολογισμού. Εγώ θα ζητήσω από τη Γραμματεία να, ζει, να, να δει όλα αυτά τα θέματα ε, που τέθηκαν. Θα μπορέσουμε να τα δούμε και με την πρόεδρο του Ινστιτούτου ε, όταν θα την έχουμε ε, μαζί μας. νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το ότι θα έχουμε κάποιον από το ΕΙΓΕ εδώ για να του θέσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα και να τα διαλευκάνουμε στο μέτρο του δυνατό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να υπενθυμίσω και εγώ αν και το είπε πολλές φορές η Φράνσις Φριτζέλαντ, 8 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι, είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Και είναι πλέον 10.35 και περνάμε στο επόμενο σημείο της τη διάταξης. Έβαλα την ώρα για το επόμενο σημείο, γιατί έχουμε μαζί μας προσκεκλημένη την Γκαμπριέλα Κουέβας, πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Μέχρι τις 11 και 4. Γι' αυτό δυστυχώς είμαι υποχρεωμένη να διακόψω τη συνεδρίασή μας μέχρι τις 11 και 4. Δυστυχώς έτσι είναι το πρόγραμμα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε νωρίτερα την προσκεκλημένη μας εδώ. Είναι σε άλλη επιτροπή του Κοινοβουλίου. Ένα καφέ θα πιούμε και τα ξαναλέμε στις 11 και 4. 1, 2. Norman Là, tu peux parler. Eh oh. Eh oh. Oh, ça m'a. Oh, oh. Non, couperez. Uh, dear members, thank you very much for your patience so far. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Η προσκεκλημένη μας θα έρθει σε λίγα λεπτά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Συνάδελφοι, έφτασε η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας στη διάρκεια αυτής της διακοπής που κάναμε. Έφτασε όμως η ώρα. Περνάμε στο σημείο 8 και έχουμε μαζί μας την κυρία Γκαμπριέλα Κουέβας Βαρών που είναι πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Όπως είπα και νωρίτερα, έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα σήμερα. Ήταν ε, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ε, εμφανίστηκε και ενώπιον της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Η κυρία Κουέβας είναι βουλευτής του Μεξικανικού Κοινοβουλίου. Θα σας πω δύο λόγια τώρα για την Διακοινοβουλευτική Ένωση. Για αυτό το όργανο, διότι Έχουμε πολλές επαφές στο τελευταίο διάστημα με διάφορους φορείς που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων. Η Διακοινοβουλική Ένωση ιδρύθηκε το 1889. Συμμετέχουν σε αυτήν τα Εθνικά Κοινοβούλια 178 χωρών. Είναι πραγματικά ένας τεράστιος οργανισμός δηλαδή. 12 περιφερειακές ε, κοινοβουλευτικές διασκέψεις ε, επίσης ε, συμμετέχουν μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η IPU είναι ένας από τους ε, ηγετικούς ε, οργανισμούς για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών, την ε, ισότητα των φύλων και την ενίσχυση της δημοκρατίας. Έχει τρεις βασικούς στόχους. Το αύξηση του αριθμού μέσω ποσοστώσεων των γυναικών που συμμετέχουν σε, βουλε... σε κοινοβούλια, υποστήριξη ε, των γυναικών στα κοινοβούλια και ε, ενίσχυση των επιτροπών που ασχολούνται με τα ζητήματα δικαιωμάτων γυναικών. Στο ε, Μεξικό, 7 και 8 Μαΐου του 2020 θα πραγματοποιηθεί το Φόρουμ για την Ισότητα μεταξύ των γενεών που αφορά και βεβαίως και την ισότητα των φίλων υπό την αιγίδα ε, του ΟΗΕ. Γι' αυτό και σας ε, ευχαριστούμε κυρία Κουέβας που είστε εδώ μαζί μας και σας δίνουμε ευθύς αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Thank you. Thank you very much for this. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική πρόσκληση. Επιτρέψτε μου να μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα, ε, στα ισπανικά δηλαδή. Πρώτα απ' όλα. Esta invitación. Me da mucho gusto poder Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται για να έρθω ε, εδώ. 130 χρόνια ε, ε, ζωής έχει η Διακοινοβουλευτική Ένωση, αλλά εγώ είμαι η δεύτερη γυναίκα μόνο που προεδρεύει αυτής της Ένωσης. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για μας και να σας πω ότι ε, Είμαι η πρώτη νέα πρόεδρος, άρα ε, γιατί εμείς λέμε ότι είμαστε νέοι μέχρι τα 45, είμαι λοιπόν και νέα και γυναίκα. Ε, η πολιτική κατάσταση δεν είναι καλή. Πρέπει να πούμε ότι ναι, μπορούμε να βελτιωθούμε και από τη διάσκεψη του Πεκίνου τα πράγματα ίσως έχουν αλλάξει και η τάση είναι θετική, αλλά πάντως... Ε, ενώ το μισό του πληθυσμού του πλανήτη είναι ε, ε, γυναίκες, μονάχα μία στις τέσσερις κοινοβουλευτικές έδρες κατέχονται από γυναίκες. Αυτό δεν είναι καλό και δεν είναι σωστό. Ε, και δεν είναι σωστό και όταν μιλάμε και για τους νέους. Ε, περισσότεροι από το 50% της του πληθυσμού του πλανήτη ε, είναι νέοι, κάτω των 30 έτη, αλλά μονάχα 2,2% των κοινοβουλευτικών εδρών βρίσκονται, κατέχονται από νέους κάτω των 30 ετών. Άρα αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό και σίγουρα σίγουρα δεν είναι δημοκρατικό. Τώρα, έχουμε πολλές στατιστικές για να δούμε ποια είναι η θέση των γυναικών στα κοινοβούλια. Ε, έχουμε κάνει δύο έρευνες, ε, είναι δύο μελέτες περισσότερο παλά ε, έρευνες. Ένα σε παγκόσμιο επίπεδο, γυναίκες δηλαδή στα κοινοβούλια και μία δεύτερη μελέτη σε περιφερειακό επίπεδο, μία ε, που αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης για τον σεξισμό ε, και για την βία κατά των ε, γυναικών στις γυναίκες και στα κοινοβούλια. Και ενώ θεωρούσαμε ότι η Ευρώπη ήταν μια ασφαλής περιοχή, Πραγματικά δεν είναι. 80% των γυναικών που συμμετείχαν είτε κοινοβουλευτικές βουλευτέ είτε ε, σχετικές με την εργασία έχουν ε, υποστεί κάποιο είδος ε, βίας λόγω του φίλου τους, ξεκινώντας από μικρά προβλήματα, φτάνοντας μέχρι την φυσική βία και την σεξουαλική παρενόχληση. Ρωτήσαμε ε, λοιπόν πώς είναι δυνατόν όταν ε, γνωρίζουν την κατάσταση οι γυναίκες να θελήσουν να μπουν στην πολιτική. Μπορεί να λέμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση, αλλά ε, εγώ πραγματικά πρέπει να σας πω ότι είμαι σαφώς υπέρ των ποσοστώσεων. Εγώ δεν νομίζω ότι ε, πολλά χρόνια σκεφτόμαστε ότι πρέπει να ε, υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ ανδρών και γυναικών για την πολιτική κατάσταση. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι επιτάχυνση της πολιτικής διαφοροποίησης έτσι ώστε να ακολουθήσουν και οι θεσμικές αλλαγές. Ε, αυτό που κάνουν οι ποσοστώσεις είναι να αλλάζουν το παράδειγμα έτσι ώστε να αλλάξει και η πολιτιστική αντιμετώπιση αντιμετώπιση. Γιατί είναι απαραίτητε οι ποσοστώσει, Μα γιατί πολλέ χώρε δεν πρόκειται να αλλάξουν ε, λόγω των καλών προθέσεων ή λόγω τη ε, απλή αδράνεια. 25 χρόνια έχουν περάσει από τη διάσκεψη του Πεκίνου και ακόμα αυτά τα στοιχεία αποτελούν ε, στοιχεία ε, πρωταρχικής σημασίας. Είπαμε ότι ναι, πρέπει κανείς, όταν θέλει κανείς να είναι politically correct, θα πρέπει να, έχει, ε, να συμπεριλάβει στην πολιτική του, στο πολιτικό του θεματολόγιο και το θέμα της των γυναικών. Αλλά δεν μπορεί να μείνουμε στα λόγια, πρέπει, χρειαζόμαστε δράσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια που εμείς σαν γυναίκες ε, ε, που βρισκόμαστε στην πολιτική ανοίγουμε τελικά δρόμους για άλλες, για τις άλλες γυναίκες και ανοίγουμε μια, ένα θεματολόγιο διεκδικήσεων και οπωσδήποτε θα πρέπει ε, η παρουσία μας και η συμμετοχή μας σε τέτοια όργανα τελικά να αντικατοπτρίζεται ή να μεταφράζεται σε, συγκεκριμένες, ε, ε, σε συγκεκριμένη νομοθεσία. Και Επομένως, όταν μιλάμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξη ε, για το 2030, θα πρέπει και εμείς ε, στα κοινοβούλια να ακολουθήσουμε την ίδια τροχιά, την ίδια διαδρομή. Ε, θα πρέπει επομένως και στην πολιτική, όταν καταρτίζονται οι πολιτικοί προϋπολογισμοί, να συνεκτιμάται πάντοτε η διάσταση των, του φύλου. Απ' την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι είναι θεμελιώδου σημασίας να χρησιμοποιήσουμε την επόμενη χρονιά γιατί οι ημερομηνίε είναι ήδη συγκεκριμένε. Όπως είπε και η πρόεδρο προηγουμένω, ε, έχουν ήδη τα Ηνωμένα Έθνη εγκρίνει μία σειρά ε, ε, συζητήσεων με την κοινωνία και έχουν τον γενικό τίτλο «Γενεά της Ισότητας». Η πρώτη διάσκεψη θα γίνει τον Μάιο 7 και 8 Μαΐου στη δικιά μου χώρα, στο Μεξικό. Και η τελευταία θα γίνει 7 με 10 ε, Ιουλίου στο Παρίσι. Μέσω αυτών ε, των ε, φόρουμ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε σε ουσιαστική αλλαγή της ποιότητας ζωής των γυναικών και αυτό πραγματικά είναι ένα σημαντικό στοιχείο της δουλειάς μας και πιστεύω ότι πολλά μπορεί να ε, πει κανείς όσον αφορά την ε, δική μας διακοινοβουλευτική ένωση που είναι μια σοβα... ένας σοβαρός οργανισμός και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ε, και στα κοινοβούλια και στα γραφεία των Υπουργών. Και αυτό που κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε στοιχεία τα οποία μας υποβάλλουν τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο σε δηλώσεις, ψηφίσματα κλπ. Ε, θα πρέπει ε, σε τούτη και στην επόμενη γενιά των γυναικών να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα ε, και εάν θέλουμε ε, να ε, επιτύχουμε την πραγματική ισότητα των γυναικών ε, θα πρέπει να περάσει ακόμα ένα αιώνας αν πηγαίνουμε με αυτόν τον ρυθμό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, κυρία Πρόεδρε, γιατί εγώ θέλω να έχουμε διάλογο που είναι κάτι πιο ζωντανό και αυτό θα ήθελα να έχω με τους παρισταμένους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Όχι μόνο για το γεγονός ότι είστε εδώ, για την παρουσίασή σας, αλλά κυρίως για την ε, δραστηριότητά σας. Γιατί βλέπουμε ότι ε, κάνετε τις, ε, τις εργασίες αυτές με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα να, να δώσω τώρα το λόγο στους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή. Η Frances Fitzgerald έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση. Να σας πω εγώ ε, για την ε, δική μου εμπειρία από την IPU. Ήμουν βουλευτής του Ιρλανδικού ε, Κοινοβουλίου τα πρώτα χρόνια της, πολιτικής, της μου δραστηριοποίησης. έλαβα γνώση της ύπαρξης αυτού του οργανισμού και συμμετείχα σε πολλές συνεδριάσεις ε, είπατε κι εσεί ότι τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια πρέπει να προσθέτουν γυναίκες στην IPU. Και θέλω να πω κι εγώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θεώρησα, βρήκα ότι ήταν εξαιρετικά διδακτική η εμπειρία μου ε, ως μέλος της αντιπολίτευσης στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο ε, το ότι είχα τη δυνατότητα να δω ποια είναι η θέση των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Ε, δεν ξέρω ε, ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχή σήμερα πια ε, γυναικών στην IPU. Φαντάζομαι ότι έχει αυξηθεί. Όμως πραγματικά πρέπει να σας πω ότι ήταν, έκανε τεράστια διαφορά στη δική μου πορεία το ότι είχα αυτή την ευκαιρία. Το ότι εκτέθηκα δηλαδή σε, αυτήν την, σε αυτό το διεθνές βήμα ως βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τις συνεδριάσεις της IPU ως εκπρόσωπος τη Ιρλανδίας. Εμείς έχουμε εισαγάγει ένα σύστημα ποσοστώσεων στην Ιρλανδία, 30% για την εκλογή ε, γυναικών, 30% ε, δηλαδή των βουλευτών θα πρέπει να είναι ε, γυναικός, γυναίκες. Το οποίο σύστημα συνοδεύεται από κυρώσεις, που είναι και το μόνο πράγμα που δουλεύει. Αυτό σημαίνει ότι αν κόμματα ε, έχουν εκλέξει βουλευτές αλλά δεν είναι το 30% εξ αυτών γυναίκες επιβάλλονται κυρώσεις οικονομικές, χρηματοδοτικές. Αν θέλουμε λοιπόν με σοβαρότητα να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό σε όλες τις χώρες. Ο μόνος τρόπος είναι οι ποσοστώσεις ως προσωρινό αναγκαστικό μέτρο, όπως λέει και ο ΙΕ, και ταυτόχρονα θα πρέπει να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, διότι το να περιμένουμε τη συνήθη διαδικασία δυστυχώς θα διαρκέσει υπερβολικά πολύ χρόνο για να δημιουργηθεί αυτή η αναγκαία κρίσιμη μάζα στις περισσότερες χώρες. Πρέπει λοιπόν να επιταχυνθούν αυτές οι δράσεις και να είναι και πολύμορφε. Και νομίζω ότι ε, στα εθνικά κοινοβούλια πολλές φορές χαράσσονται πολιτικές οι οποίες είναι αρκετά ε, ε, επιθετικές. Ε, υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο ε, σχετίζεται με τη δημοκρατία το οποίο δυστυχώς μας υπάρχουν διάφορα προβλήματα που απειλούν ακόμη και την ίδια την ύπαρξη της δημοκρατίας. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν γυναίκες. Ευχαριστώ η κυρία Νόιχλ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Εγώ ε, είμαι ευρωβουλευτής από τη Γερμανία. Στο δικό μου κόμμα έχουμε εισαγάγει ποσόστοση και έχουμε και ένα σύστημα φερμουάρ, το οποίο λέει δηλαδή ότι θα πρέπει εναλλάξ να υπάρχουν ένας άντρας, μια γυναίκα. Έτσι καταρτίζονται οι, ε, τα, τα ψηφοδέλτια. Ε, αυτό βεβαίως δεν ε, εξάλληψε το φαινόμενο να εκλέγονται πολλοί άντρες. Ε, γι' αυτό και εμείς ε, έχουμε απομακρυνθεί λίγο από την έννοια της ποσόστοσης και οδηγούμαστε πιο πολύ στην, ε, στην έννοια της ισοτιμίας. Διότι πρέπει να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα. Ε, υπάρχει μια κατανομή, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράδειγμα, ανα, ε, κατά χώρε ανάλογα με τον πληθυσμό των χωρών. Όμως ε, δεν υπάρχει σχετική κατανομή όσον αφορά τις γυναίκες. Γι' αυτό και εμείς απαιτούμε ότι ε, μια περιφερειακή, ε, ε, ακόμη και εντό των κρατηδίων της Γερμανίας, ποσόστοση δεν θα πρέπει ποτέ να είναι αυστηρότερη από μια αντίστοιχη ποσόστοση για τις γυναίκες. Και να υπάρχουν και συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες να μπορούν να καταλαμβάνονται μόνο από γυναίκες. Τέλος, η ποσόστοση είναι ένα εναρκτήριο μέτρο αν θέλετε η ισοτιμία είναι η ισότητα που αφορά την, την, την άφηξη, το τέλος δηλαδή. Ε, δεν είναι ένα εναρκτήριο μέτρο. Διότι ανάμεσα στις ε, εκλογικές διαδικασίες και στην κατάληψη θέσεων Τελικά κάτι πάντοτε συμβαίνει και είναι περισσότεροι οι άντρε αυτοί που έχουν, κατέχουν τι υψηλέ σημαντικέ θέσει. Γι' αυτό και κάτι πρέπει να κάνουμε. Καλή υποσώστοση όμως όμω θα πρέπει να δοθεί ε, ιδιαίτερη έμφαση και στην έννοια τη ισοτιμία όσον αφορά τι θέσει που θα καταλαμβάνονται. Ευχαριστώ, η κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και για τις προσπάθειες που καταβάλλετε. Ισοτιμία ανδρών και γυναικών είναι βεβαίω ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί σε όλου του τομεί και σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, με ενοχλεί ιδιαίτερω και το εκφράζω ε, σφοδρότατα, η έννοια τη ποσόστοση. Αν ε, ε, λέτε εσεί μάλλον το επιχείρημα ότι το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι γυναίκες, αλλά μόλις το 25% των βουλευτών σε όλο τον κόσμο είναι γυναίκες. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια ε, εσφαλμένη βάση επί τη οποίας θέλετε να θεμελιώσετε την ανάγκη για την, για την θέσπιση ποσόστοσης. Διότι υπάρχει μια, ε, ε μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε απλά να την αγνοήσουμε. Οι λιγότερες γυναίκες ε, ενδιαφέρονται για την πολιτική. Μπορεί κανείς να διαμαρτύρεται, να ενοχλείται από αυτή την πραγματικότητα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό και πραγματικά ε, ε, για να ε, καταλήξουμε σε έναν ε, τέτοιο στόχο θα πρέπει ενδεχομένω ακόμη και να αναγκαστούν γυναίκες να ασχοληθούν με πράγματα τα οποία δεν τι ενδιαφέρουν. Γι' αυτό και βρίσκω πολύ προβληματική την έννοια της ποσόστοσης. Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά παραβίαση του ε, ε, ε, του ελεύθερου δικαιώματος του εκλέγην. Η θέσπιση λοιπόν ποσόσως για τις γυναίκες, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί και μια αντανάκλαση ε, του σεξισμού που πράγματι υπάρχει. Ενδεχομένως το αντεστραμμένο του είδωλο, αλλά ε, είναι γεγονός ότι, ε, γιατί είναι σαν να λες ότι οι γυναίκες δεν μπορούν από μόνες τους, με τις ίδιες τους τις δυνάμεις, να κατακτήσουν τέτοιες σημαντικές θέσεις, αλλά θα πρέπει να τις βοηθήσουμε και να τις... Ε, ε, να συμβάλλουμε κι εμείς με θεσμικά μέτρα. Εγώ ε, είμαι πολύ περήφανη που μπορώ για τον εαυτό μου να πω ότι κατάφερα όσα κατάφερα γιατί είμαι μια δυνατή γυναίκα, μια αποφασιστική γυναίκα. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι ένας ε, σεξισμός ε, από την ανάποδη η ποσόστοση και εκφράζω την ε, διαφωνία μου. Ευχαριστώ η κυρία Ραφαέλα. Thank you. Um, thank you for your Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την παρουσίαση και την παρουσίαση, παρουσία σας. Το περασμένο μήνα δημοσιεύτηκε μια εξαιρετική έκθεση για τον σεξισμό, την παρενόχληση και τη βία τα κοινοβούλια της Ευρώπης και μερικά από τα στοιχεία πραγματικά σοκάρουν. Δείχνουν ότι 85,2% γυναικών βουλευτών έχουν υποστεί ψυχολογική παρενόχληση κατά τη διάρκεια τη εξάσκηση των καθηκόντων του. 46,9% έχουν λάβει απειλέ θανάτου ή, θανα... ξυλοδαρμού. 24,7% σεξουαλική βία και 67,9% ήταν στόχο σχολείων για την, σωματική τους, την εξωτερική τους εμφάνιση βάσει των στερεοτύπων. Η έκθεση δείχνει ότι κυρίως οι νεαρές βουλευτίνες, αυτές που εργάζονται για τα γυναικεία δικαιώματα, είναι ευκολότερο στόχο. Προσωπικά ανησυχώ πολύ. Και εγώ έχω υποστεί διάφορα, όπως κι άλλες γυναίκες φαντάζομαι εδώ, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα και κυρίως από τότε που είμαι βουλευτής εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για ισχυρή εκπροσώπηση στα πλαίσια του Κοινοβουλίου εδώ τουλάχιστον και ίσως θα μπορούσατε να πείτε περισσότερα ιδίω για το τι πορίσματα έχετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι πιστεύετε ότι έχει κάνει ως τώρα η διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Έχει κάνει αρκετά. Τι περισσότερο θα μπορούσε να γίνει. κυρία Jones. Ε, θα μιλήσω αγγλικά μια και είμαστε ακόμα εδώ. <laughs> Μετά την τρίτη μέρα του Brexit. Πολύ ευχαριστούμε που ήρθατε και συγχαρητήρια για το διορισμό σας, την εκλογή σας τέλο πάντων. Είναι πολύ καλό που μια γυναίκα γιατί μιλά για τα δικαιώματα των φίλων και την ισότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν κάποιες μελέτες για τις συνοβουλευτικές έδρες. Εγώ εκπροσωπώ την Ουαλία 40 έδρες έχουμε στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκπροσωπώ τους εργατικούς. Και έχουμε το λεγόμενο σύστημα φερμουάρε, όπως το λέμε στην Αγγλία, και έχουμε και ποσοστώσεις. Ε, υπήρχαν βέβαια κάποιες έντρες που δεν καλύπτονταν από αυτή την δυνατότητα και ποτέ δεν επέλεγε μια γυναίκα για να τις καλύψει στους καταλόγους των ε, καλύτερων υποψηφίων, εκτός από δύο φορές που έγιναν τις συγκεκριμένες εκλογές. Ε, στα εκατοντάδες χρόνια λειτουργίας ε, των εκλογών στην Ουαλία δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Τα ανοιχτά ψηφοδέλτια λοιπόν δεν επιτρέπουν στις γυναίκες βουλευτές, βουλευτίνες να κάνουν κάτι και είμαι βέβαιη ότι αυτό συμβαίνει και αλλού και όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σίγουρα και σε άλλες χώρες. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν, λαμβάνοντα αφορμή από τα σχόλια τη συναδέλφου. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω διαβάσει ακόμα την έκθεσή σα. Θα το κάνω όμω. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει ένα συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, λόγω χάρη κάποιο παράπτωμα για την ε, βία κατά των γυναικών πολιτών. Ή τουλάχιστον να είναι ένα στοιχείο που επιβαρύνει τη θέση του κατηγορουμένου σε οποιαδήποτε εκδίκαση υπόθεση. Δηλαδή να έχει και αυστηρότερη ποινή. Αυτά ως προς τις κυρώσεις και την ποσόστοση. Αλλά η ισότητα στις ευκαιρίες είναι ένα πράγμα. Το θέμα είναι ότι γίνεται και με το αποτέλεσμα. Γι' αυτό μιλάμε για την εξισορρόπηση των δύο φύλων και όχι μόνο για ισότητα. Και μετά ε, μιλάμε για ε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ψηφοφόρους μας, υποτίθεται. Εάν οι ψηφοφόροι μας είναι κάτω των 30 είναι ανάπηροι, έχουν οποιοδήποτε θέμα, ε, είναι ε, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κατηγορία πρέπει να εκπροσωπούνται. Οπότε είναι λογικό να εκπροσωπούνται και γυναίκε, όχι μόνο οι άντρε. Και τέλος μια έκκληση. Να χρησιμοποιούμε το σύστημα ΣΥΝΤΟ περισσότερο στη δουλειά μας. Δεν ξέρω αν το κάνουμε αυτό, αλλά τουλάχιστον έχουμε έτσι ένα αποτύπωμα του τι γίνεται. Πριν από 40 χρόνια πέρασε αυτή, εγκρίθηκε αυτό το εργαλείο. Ό,τι λοιπόν μας προσφέρει το σύστημα αυτό πρέπει να το αξιοποιούμε, όπως η κατάλογη υποψηφίων ε, βάσει του ΣΥΝΤΟ. για να υπάρχουν γυναίκες οπωσδήποτε στις, ε, στους καταλόγους των ε, υποψηφίων τουλάχιστον από την πλευρά των εργατικών θα γίνει αυτό μέχρι να φτάσουμε την πραγματική ε, εξισορρόπηση, ε, όχι απλώς ε, την ισότητα. Να χρησιμοποιούμε λοιπόν το σύντο στις εργασίες μας. Ευχαριστούμε. Κυρία Μελό. Η κυρία Κραβάισκα και μετά κλείνω το κατάλογο των αγοριτών. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και βλέπω ότι θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε κιόλα. Ναι, ευχαριστώ να σχολιάσω από αυτό που μόλις είπε η συνάδελφος στην ίδια σειρά. Εγώ δεν είμαι φοβερή φαν των ποσοστώσεων, αλλά κάποιοι νομίζουν ότι είναι η τέλεια συνταγή και απειλείονται έτσι όλα τα προβλήματα για την έλλειψη γυναικείας εκπροσώπησης στην πολιτική. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι η απουσία γυναικών στην πολιτική δεν έχει να κάνει με το ότι δεν ενδιαφέρονται για τα πολιτικά προβλήματα, για τα δικαιώματα των πολιτών είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά πρότυπα το πρόβλημα και οικονομικοί περιορισμοί επίσης προβάλλονται την ε, συμμετοχή τους. Η κουλτούρα μας, η νοτροπία μας και η νοτροπία που επικρατεί στα πολιτικά κόμματα επίσης είναι ένα πρόβλημα για τις γυναίκες, καθώς και οι ώρες εργασίας πολλών ε, πολιτικών θεσμικών οργάνων δεν είναι φιλικές προς τις υποχρεώσεις που έχουν οι γυναίκες, ιδίως οι νεαρές που μπορεί να έχουν και παιδιά. Πρέπει να φροντίσουν και τις οικογένειές τους και θα πρέπει να προσπαθήσουν να συνδυάσουν και τα δύο. Ήταν δύσκολο ας πούμε να κανονίσουμε διαφορετικά τις ώρες εργασίας για μένα που υπήρξα βουλευτής και έπρεπε να πάω το ωράριο της ε, καθημερινότητας από τις 2.30 μέχρι τα μεσάνυχτα για να μπορέσω να έχω χρόνο. Πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τα παιδιά του. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι συμβαίνει γενικότερα στην κοινωνία με την πολιτική. Γιατί είναι ωραίο που έχουμε αυτή τη συζήτηση εδώ σε αυτή την αίθουσα. Λε και δεν συμβαίνει τίποτα απ' έξω. Εγώ πάντως πρέπει να πω ότι εκεί που εργαζόμουν σε μια εφοπλιστική εταιρεία εμ, ε, υπήρχαν τα ίδια προβλήματα, όπως και εδώ, και γενικά αυτά συμβαίνουν σε ολόκληρη την κοινωνία. Στη Βόρεια Ιρλανδία, λοιπόν, σίγουρα από τους υποψηφίου μας 10 θα είναι γυναίκες. Εγώ είμαι ε, ηγέτης του κόμματος ως γυναίκα. Έχουμε διαφορετική ε, κουλτούρα. Θα κατεβάσουμε οπωσδήποτε τις 10 αυτές γυναίκες ως υποψηφίου και μπορεί κανείς να διοργανωθεί διαφορετικά. Είναι κρίσιμη σημασία σε αυτό όπως και να έχουμε στόχου, όπω ποσοστώσεις των αριθμών των γυναικών που θέλουμε. Πρέπει για να υπάρχει επιλογή, η δυνατότητα επιλογής γυναικών από τα θεσμικά όργανα να φτάσουν οι γυναίκες ω εκεί. Δεν είναι ότι του λείπουν τα ταλέντα ή των ενδιαφέρον. Είναι άλλα τα προβλήματα. Το μόνο άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι η επιγραμμική παρενόχληση, η παρενόχληση στο ίντερνετ. Είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και έχει στόχο κυρίως τις γυναίκες. Πολύ συχνά εγώ η ίδια έχω δεχτεί, όπως και άλλες, απειλές, ε, σωματικές, ε, φραστικές και πολλές φορές και στο γραφείο μου μέχρι ε, και εκεί. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν μπορεί να γίνει ένα επιβραντικό στοιχείο, αλλά οποιαδήποτε προσβολή κατά των πολιτικών θα έπρεπε να είναι επιβραντικό στοιχείο. Δεν είναι απλώ προσβολή ενό δημοσίου προσώπου, είναι προσβολή ενό λειτουργήματο και του δημοκρατικού συστήματο. Όλοι οι πολιτικοί αξίζουν να προστατεύονται από τέτοιου είδου σωματικέ και φραστικέ απειλέ στο διαδίκτυο. Πρέπει η κοινωνία να λειτουργεί λίγο πιο ε, ομαλά και το μποϊκοτάζ δείχνει ότι πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα που επικρατεί, η νοοτροπία στα διάφορα θεσμικά όργανα και τις οργανώσεις. Δηλαδή, γυναίκε να μην εκλέγονται βάσει ποσοστώσεων και μετά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με το λειτουργήμα που του ανατέθηκε να το συνδυάσουν με την υπόλοιπη ζωή του εκτό λειτουργήματο. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο δράση και να αλλάξει η κουλτούρα που επικρατεί στον χώρο τη πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ. Ελιζαμπέτ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Στην Πολωνία έχουμε νομοθεσία που προβλέπει ότι στα ψηφοδέλτια για τις εθνικές εκλογές πρέπει να, για τις κοινοβουλευτικές εκλογές πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 45% γυναικών. Το 2016 είχαμε 25% γυναίκες και τις τελευταίες εκλογές 43,3%. Βλέπετε να υπάρχει αύξηση στην εκπροσώπηση γυναικών στα ψηφοδέλτια ε, στις εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές. Όμως είναι εξίσου αλήθεια και θα συμφωνήσω εδώ με αυτό που είπε η κυρία ότι οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την συμμετοχή τους στην πολιτική. Αυτό αντικατοπτρίζεται και από την συμμετοχή του σε πολιτικά κόμματα. Εάν δείτε τη σύνθεση των πολιτικών κομμάτων, το 20-30% μόνον είναι γυναίκες. Και όταν συζητώ μαζί τους, το λένε και έξω τα δόντια. Δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει στην πολιτική που είναι τόσο επιθετικά τα πράγματα, που χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και γλώσσα, που διαρκώς ε, τους... Ε, τις αντιμετωπίζουν με συγκεκριμένα στερεότυπα. Οι γυναίκες λοιπόν δεν έλκονται από την πολιτική όπως από άλλους τομείς της ζωής. Ε, Πρέπει να είναι διαρκώς παρούσα στο πολιτικό βίο για να εκλέγονται και να εκπροσωπούνται στα κοινοβούλια. Εγώ είμαι πολιτικός εδώ και πέντε χρόνια και ασχολούμαι με τα θέματα αυτά στην αρχή. Κατέβηκα σε ένα κύκλο που υπήρχαν μόνο άντρες. Εξελέγησα σε τοπικό επίπεδο. Και βεβαίως θέλουμε να μπούμε στη Βουλή, όχι γιατί είμαστε νέε ή μεγαλύτερε, όμορφε ή άσχημε, αλλά γιατί έχουμε πράγματα να προσφέρουμε, έχουμε κάτι να κάνουμε και πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό απαιτείται νομοθεσία. Εμείς στην Πολωνία την έχουμε. Αλλά δεν είναι ε, τέλεια ε, η συνταγή της ε, επίλυσης όλων των προβλημάτων. Δεν είναι πανάκια. Πρέπει λοιπόν να βρούμε πώς θα σώσουμε, πώς θα βοηθήσουμε τους αυτούς μας. Θα επικεντρωνόμαστε διαρκώς στο φίλο μας και στη διάσταση αυτή ή στο τι μπορούμε να προσφέρουμε, διότι νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην πολιτική. Και το λέω και για την Πολωνία. Τα πράγματα αλλάζουν προ το καλύτερο. Δείτε τι τελευταίε εκλογέ ε, στην Πολωνία και τι εθνικέ κοινοβουλευτικέ και τι εκλογέ Και τι τοπικέ. Είδαμε να συμμετέχουν και να εκλέγονται πολύ περισσότερε γυναίκε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Πολύ γρήγορα, ένα λεπτό, η Ρεν Αλλά παρακαλώ γρήγορα για να έχει την ευκαιρία καλεσμένη μα απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα όντω. Στη Γαλλία έχουμε ε, πολλές, ε, ε, πολλούς νόμους όσον αφορά τις εκλογικές διαδικασίες. Μία, ένας νόμος είναι του 2015, βάσει της οποίας αντί να ψηφίζουμε για μία θέση, ψηφίζουμε για ένα ζευγάρι ε, και αυτό ε, έδωσε την ε, δυνατότητα να βάλουμε καινούρια πρόσωπα στην πολιτική, μια και πολλές γυναίκες, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, θεωρούσαν ότι δεν είχαν θέση, δεν μπορούσαν να μπουν στην πολιτική. ναι, υπάρχουν επίσης αυτοί οι κατάλογοι εκλογικοί που εμείς τους λέμε σαμπαντά, που είναι δηλαδή ένας άνδρας, μία γυναίκα. Ε, και επομένως καταλαβαίνετε ότι γίνονται πολλές προσπάθειες νομίζω ότι αυτό το θέμα του ζευγαριού είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ε, υπάρχει αυτό το σύστημα φερμουάρα, ας πούμε, και στην ε, Ιταλία, αλλά μετά ε, δεν έχει εκλογικό αποτέλεσμα με την έννοια ότι εκλέγονται περισσότεροι άνδρες από γυναίκες. Όσον αφορά την κατάχρηση ή την κακή συμπεριφορά κατά των γυναικών πολιτικών, πραγματικά είναι κάτι απαράδεκτο. Νομίζω ότι η μόνη κριτική που θα έπρεπε να γίνεται εναντίον μας ε, θα πρέπει να αφορά το έργο μας ε, και τις ικανότητές μας ε, γιατί είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση να βαλόμεθα από παντού. Ευχαριστώ πολύ. Ε, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Κουέβο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Ε, νομίζω ότι και από αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί εγώ συμφωνώ και υποστηρίζω τις ποσοστώσεις. Εγώ ε, ε, ήμουν 21 ε, ετών όταν πρωτομπήκα στο κοινοβούλιο της χώρας μου και τότε δεν υπήρχαν ούτε ποσοστώσεις ούτε τίποτα. Ούτε για γυναίκες, ούτε για νέους, ούτε... και με μπήκα λοιπόν σε μια βουλή 500 ατόμων. Ήμουν τοπική βουλευτής, εκλέγηκα χωρίς καμία ποσόστοση. Και στις δημοτικές εκλογές ε, επί 16 περιφερειών ε, Ήμουνα η μοναδική γυναίκα δήμαρχος. Μετά ξαναέγινα, φανταστείτε, σε μια, χώρα τόσο, σε μια πόλη τόσων εκατομμυρίων, στην πόλη του Μεξικό, εν μια γυναίκα δήμαρχος. Και μετά ξαναέγινα έγινα ε, γερουσιαστής και μετά βουλευτής. Σε καμία περίπτωση δεν ε, πήρα τη θέση που πήρα λόγω των ποσοστώσεων ε, για τις γυναίκες. Και στις πρεσινές εκλογές εγώ ήθελα να είμαι υποψήφια στη δικιά μου περιφέρεια. Ε, και δεν μπόρεσα να είμαι υποψήφια στην δικιά μου ε, ε, περιφέρεια γιατί είχαμε πλέον ποσοστώσεις και στην δικιά μου περιφέρεια έπρεπε να παρουσιαστούν μονάχα υποψήφοι άντρες. Ε, γιατί πλέον υπάρχει το σύστημα των ε, ποσοστώσεων. Επομένως, εγώ, αντί να βελτιώσω την κατάστασή μου ε, βάσει των ποσοστώσεων φύλου, εγώ είχα χειρότερη αντιμετώπιση. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως Κανένας μέχρι τώρα δεν έχει πει, στη διάρκεια των αιώνων, ε, δεν έχει πει εάν ε, έχουν περισσότερο ψηλότερο IQ ε, οι άνδρες από τις γυναίκες ή αν έχουν περισσότερα προσόντα οι άνδρες από τις γυναίκες. Ποτέ δεν έγινε μια τέτοια μελέτη και δεν έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Επομένως αυτά πρέπει να τα βγάλετε από το μυαλό σας. Ustedes Εσείς μιλήσατε για άλλα θέματα για τον, ο, ο τρόπος πολιτικής, ο τρόπος του πολιτεύεστε, ε, η γλώσσα της πολιτικής, όλα αυτά τα έχουν διαμορφώσει οι άνδρες και ακόμα και σε άλλους τομείς, τεχνικούς τομείς, τεχνικά παιδεία, χρηματοοικονομικά κτλ. Ακόμα εξακολουθούν οι άνδρες να έχουν ε, την μαζική παρουσία και όχι οι γυναίκες. Επομένως, λέω, ποσοστώσεις ναι, όχι για πάντα, αλλά για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πολιτιστική αλλαγή. Ναι, τώρα μιλάμε λόγω συγκυρίας ε, μιλάμε πολύ για ε, γυναικεία ζητήματα, για τις γυναίκες και τα λοιπά, αλλά όταν θέλουμε να μεταφράσουμε τα ε, λόγια σε έργα και σε πράξεις, τότε επιβραδύνεται τρομερά η διαδικασία. η αύξηση των, της συμμετοχής των γυναικών πέρσι ήταν 0,9% ε, και τον προηγούμενο χρόνο 0,1. Ε, με, αυτήν την, ε, με αυτό το ρυθμό θα χρειαστούμε 250 χρόνια μέχρι να επιτύχουμε την ισότητα των φύλων στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και νομίζω ότι είναι εύγλωτη αυτή η αριθμή. Όταν αναφερόμαστε στην ε, βία που υφιστάμεθα εμείς οι γυναίκες στην πολιτική αφορά και τον τρόπο συμπεριφοράς ε, και ε, τον λόγο και τα λοιπά και τις πράξεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς θέλουμε να διώξουμε τους άντρες. Όχι. Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει μαζί με τους άντρες γιατί διαφορετικά θα συνεχίσει η βία κατά των γυναικών. Χρειαζόμαστε μία ε, συνολική ε, συμπεριληπτική αλλαγή ε, έτσι ώστε να αλλάξουν πραγματικά οι νοοτροπίες και εάν δεν αλλάξουμε τους ε, κανόνες δεν θα αλλάξουν και τα κίνητρα ε, που μπορεί να δώσουν οι ηγεσίες των διαφόρων κομμάτων έτσι ώστε να προωθήσουν γυναικείες ε, φιγούρες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες που θα πυροδοτήσουν την αλλαγή. Και ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν κοινωνίες ε, οι οποίες ε, έχουν μεγαλώσει τους άνδρες και τις γυναίκες ε, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένο πολιτισμό, κοινωνίες οι οποίες είναι ανδροκυριαρχούμενες, δεν έχουν κανένα λόγο να αλλάξουν γιατί δεν έχουν μάθει ότι υπάρχει ένα άλλο μοντέλο και επομένως αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να μάθουμε να αλλάζουμε τα ε, υποδείγματα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οικοσυστήματα με δικτύωση που θα δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες που είναι νέες ε, να αλλάξουν την οτροπία τους. Οι γυναίκες οι οποίες μαθαίνουν από μικρές ότι θα πρέπει να μεγαλώσουν, να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά ε, και όχι κάτι άλλο. Πώς σε αυτές τις γυναίκες να τους εμφυσίσουμε την αγάπη για άλλες για άλλες δραστηριότητες δεν υπάρχουν οι υποδομές ε, για τις ε, γυναίκες ε, να μπορέσουν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν και όλες οι υποδομές που πρέπει έτσι ώστε να τις βοηθήσουν να μπορέσουν να είναι και πολιτικοί και γυναίκες. Λίγες είναι οι, λίγα είναι τα κοινοβούλια τα οποία έχουν και παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγία κλπ. Εν πάση περιπτώσει πώς, αν δούμε πώς αυξήθηκε η συμμετοχή των γυναικών τα τελευταία 25 χρόνια στα κοινοβούλια και πώς τροποποιούνται οι δίκτυες ανάπτυξης για τις γυναίκες, βλέπει κανείς ότι δεν ε, ε, διαπιστώνεται καμία ε, σημαντική βελτίωση, ότι οι ε, παρουσία, η μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στα κοινοβούλια έχει οδηγήσει σε ε, τροποποίηση των ρυθμών ανάπτυξης. Επομένως θα πρέπει να αναπτύξουμε και αυτή είναι την θεματολογία ε, που είναι συνδεδεμένη με το φύλλο όχι μόνο στα κοινοβούλια αλλά και μέσα στην κοινωνία. Ε, πολιτική βία ε, κατά των γυναικών. Ε, χαίρομαι που αναφερθήκατε σε αυτήν την μελέτη που κάναμε μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ τρομακτικά αυτά που είδαμε το Συμβούλιο της Ευρώπης μαζί με τη Διακοβουλευτική Συνέλευση ξεκίνησε μια εκστρατεία με τίτλο Not in my Parliament, όχι στο δικό μου κοινοβούλιο, ε, έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση. Και επίσης ε, εμείς αυτή τη στιγμή διαμορφώνουμε διάφορα εγχειρίδια ε, σχετικά με το ας πούμε ποιοι κανόνες πρέπει να υπάρχουν, κώδικα συμπεριφοράς, κώδικας ακόμα και κυρώσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια καλή στρατηγική. Ειλικρινά, δεν πιστεύω έχουμε μία νομοθεσία, έχουμε νόμο κατά της πολιτικής βίας κατά των γυναικών. Ε, αλλά στις τελευταίες εκστρατείες υποτίθεται ότι εφαρμόστηκε στο Μεξικό. Αλλά ε, πραγματικά... Ε, εν τέλει αυτό το βλέπει άσχημα η κοινωνία αρνητικά γιατί λέει και γιατί εσένα να σε προστατέψουμε περισσότερο από ό,τι άλλους. Νομίζω ότι σε σχέση με το ε, κίνημα Me το πιο σημαντικό του στοιχείο ήταν ότι έμαθε στις γυναίκες να καταγγέλουν, έμαθε στις γυναίκες να καταλαβαίνουν, ε, να ε, έχουν συνείδηση του ότι αυτού του είδους η παρενόχληση δεν είναι κάτι φυσιολογικό δεν είναι κάτι σωστό, δεν είναι κάτι που πρέπει να υφίστανται και επομένως πρέπει να καταγγέλουν. Επομένως πρέπει να είναι σαφές ότι οποιαδήποτε εκδήλωση βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να ε, τιμωρείται. Προσπαθώ τώρα να καλύψω και όλες τις ερωτήσεις που υποβάλλατε και τα σχόλια που κάνατε όσον αφορά τις ε, ποσοστώσεις. Ε, να σας πω ότι στις μελέτες που έχουμε σαν ε, Ένωση, Κοινοβουλευτική Ένωση, υπάρχει κάτι που λειτουργήσε καλά. Πρώτον, ότι ναι, υπάρχουν ποσοστώσεις στη δικιά μας οργάνωση, όπως το είπε η κυρία Φιτζέραντ. Και ξεκινήσαμε λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχουν αντιπροσωπείες όπου ε, αν δεν υπήρχε ισότητα, τουλάχιστον ε, ισότητα εκπροσώπησης, τουλάχιστον υπάρχει κάποια εκπροσώπηση ε, γυναικών. Ε, δεν το κάναμε αμέσως, αλλά τώρα πλέον όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείες έχουν γυναίκες. Ίσως μία-δύο δεν έχουν καθόλου. Επίσης, ξεκινήσαμε κάποια μέτρα για τους νέους κοινοβουλευτικούς και στην τελευταία μας συνεδρίαση, στην τελευταία θητεία μάλλον, αρχίσαμε να επιβάλλουμε τιμωρίες, κυρώσεις στα πολιτικά κόμματα που δεν ε, περιλάμβαναν γυναίκες στις αντιπροσωπείες τους. Να σας πω ότι από τις 10 χώρες με μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στα κοινοβούλια, 8 από αυτές τις 10 χώρες είναι γιατί έχουν ποσοστώσεις. Ε, οι άλλες είναι η Ρουάντα, αυτό εξηγείται από τη γενοκτονία, ε, και η Κούβα που εξηγείται από την παρουσία των γυναικών ε, από, στη διάρκεια της Επανάστασης. Όλες οι άλλες έχουν ε, ποσοστώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, να επιταχυνθεί η πολιτιστική αλλαγή. Ε, εάν, εάν σήμερα περισσότερο από ποτέ δεν πείσουμε τις γυναίκες ότι η θέση τους δεν είναι στο σπίτι, δεν θα κάνουμε τίποτα. <clears throat> Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ε, herzlichen Dank. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Θεωρούμε ότι η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ένα εξαιρετικό βήμα από το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτήν την πολιτιστική και πολιτισμική μεταστροφή που βρίσκεται ε, σε εξέλιξη και χαιρόμαστε πάρα πολύ για το έργο που θα γίνει έως την συνδιάσκεψη του Μαΐου στο Μεξικό. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτού του σημείου της ημέρας της διάταξης και κηρύσω τη λήξη της ε, συνεδρίασης της Επιτροπής μας και ε, κηρύσω ευθύ αμέσω την έναρξη τη κοινή συνεδρίασης που θα γίνει με την Επιτροπή Ανάπτυξη. Το φως θα το ξανανάψουμε. Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμη για σήμερα. <laughs>